Przewodniczący! E, Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ να καθίσετε. Otwieram posiedzenie przerwane Λοιπόν, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης που είχε αρθεί την προηγούμενη φορά στο Στρασβούργο. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνόδου υπάρχουν στους φακέλους σας. Μήπως υπάρχει κανένα σχόλιο επ' αυτόν η παρατήρηση, όχι, εγκρίνονται. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Την Δευτέρα επλήγει η Ουγγαρία από τη χειρότερη θεομηνία της ιστορίας της. Δηλαδή τοξικά οι γράδι έφυγαν... από μία αποθήκη. Υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες. Θα ήθελα λοιπόν να στείλουμε τηλεγραφήματα συλληπιτήρια εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να σας πω ότι αύριο θα γιορτάσουμε, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας της Άννας Πολιτικόσκαγια που όπως ξέρετε είχε δώσει τη ζωή της για να ανακαλύψει την αλήθεια για αυτά που συνέβαιναν στον Κάφκασο στην Τσετσενία. Έχουμε από τη φόρο τιμή στη μνήμη της κυρίας Πολικόφσκα για στον αγώνα της για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης αφού δώσαμε το όνομά της σε μία από τις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν ξεχνούμε ούτε άλλους δολοφονηθέντες δημοσιογράφους, την κυρία Αναταλία Εστεμίροβα και την κυρία Αναστασία Μαρμούροβα καθώς και άλλους αγωνιστές νομομαθείς όπως τον κύριο Στανισλάβ Μαρκελόφ, Σεργέη Μανίτκι και άλλους. Οι συνθήκες της δολοφονίας τους δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί και ζητούμε από τις ρωσικές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να σεβαστούν τις αρχές του κράτους δικαίου και να τερματίσουν επιτέλους αυτή την κατάσταση αβεβαιότητας. Στις 10 Οκτωβρίου θα εορτάσουμε την Διεθνή ημέρα κατάργησης θανατικής ποινής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να οργανώσει όπου μπορεί σε όλες τις χώρες ένα μορατόριο κατά της θανατικής ποινής. Δεν μπορεί να θεωρηθεί η θανάτωση ως καταδίκη νόμιμη βλέπουμε ότι και στη Ρωσία, στον Μπουρούντι και στο Τονγκό γίνονται κινήσεις για την κατάργησή της. Δυστυχώς όμως στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ιαπωνία εφαρμόζονται ακόμη θανατικές εκτελέσεις. Φρονούμε ότι η δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, αλλά αυτό που μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι ο αριθμός των εκτελέσεων που συμβαίνουν σε χώρες όπως η Κίνα ή το Ιράν ζητούμε από τις αρχές των χωρών αυτών να τερματίσουν την πρακτική αυτή. Κυρίες και κύριοι, έλαβα από την ομάδα του ΕΛΚ αιτήματα ορισμού μελών ορισμένων αντιπροσωπείων Εάν δεν ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα εγκριθούν οι ορισμοί αυτοί. Και τώρα κυρίες και κύριοι περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Σήμερα και αύριο με σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων θα προτείνω τις εξής αλλαγές. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες είναι υπέρ των αλλαγών αυτών. Λοιπόν, ειδού την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, θα προσθεθεί στην μέση διάταξη ένα νέο σημείο η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις κοινωνικές ρήτρε της ε, συνθήκης της Λισαβόνας μετά από, μετά από τη συζήτηση για τη βιοπικιλότητα. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε για την διαγραφή της προφορικής ερώτησης για τα εμπορματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα και την πέμπτη να αρχίσουν οι ψηφοφορίες στις 11.30 αντί στις 11 και την Πέμπτη επίσης να διαγραφεί η συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Μάνικα ως προς τον διορθωτικό προπολογισμό 2-2010 διότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει και επομένω δεν υπάρχει λόγος να γίνει η συζήτηση αυτή αύριο. Τώρα, ως προς αυτό που σας είπα για σήμερα, για τα εμπορευματοκιβώτια, μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε. Ο κύριος Βόρτμαν Κόλ έχει ήδη ζητήσει το λόγο. Η κυρία, κυρία. Κύριε Πρόεδρε, το ΕΛΚ πάντοτε δέχεται συζήτηση για κοινωνικά θέματα στις Ολομέλειες. Πρέπει όμως οι συζητήσεις αυτές να είναι σωστά προετοιμασμένες και γι' αυτόν τον λόγο στη διάσκεψη των Προέδρων είχε αρχικά αποφασιστεί η πρόταση της ομάδας των σοσιαλιστών να γίνει συζήτηση για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και τις κοινωνικές ρήτρες της Λισαβόνας είχε αποφασιστεί η συζήτηση αυτή να γίνει μια πλειοψηφία το είχε δεχτεί αλλά πρώτα να γίνει στην Κοινωνική Επιτροπή. Αυτό φρονούμε και σήμερα, γιατί το θέμα είναι δύσκολο και πολύπλοκο. Οι φιλελεύθεροι έχουν εδώ μεταξύ αλλάξει στάση και θέλουμε η συζήτηση προηγουμένως να γίνει στην Κοινωνική Επιτροπή. Ακριβώς γιατί το θέμα είναι πολύπλοκο. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προσκόμματα, αλλά εμείς θα απόσχουμε κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της συζήτησης αυτής. Ευχαριστούμε για την εξήγηση αυτή, κυρία μου. Συμπεραίνω λοιπόν ότι το σημείο αυτό που ζητιέται να θα μπει στη σημερινή, σημερινή διάταξη ακόμα και αν απέχει η ομάδα του ΕΛΚ, γιατί οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες έχουν εγκρίνει την προσθήκη. Άλλες δηλώσεις ή σχόλια, δεν βλέπω. Επομένως, εγκρίνεται έτσι με αυτές τις ανθρωποποιήσεις η ημερήσια διάταξη. Στις 3.30 θα γίνει η πανηγυρική συνεδρίαση με τον πρόεδρο του Ανατολικού Τιμόρ. Θα ήθελα λοιπόν σε 20 λεπτά να είστε έτοιμοι να επιστρέψετε εδώ. Σε 20 λεπτά, ακριβώς σε 20 λεπτά στις 3 και 30 άκρη.